μέσα Φέρμπερ χρηματοπιστωτικά μέσα κατά χρήση αρβορών και κανονισμός. Έχετε τον λόγο κύριε Φέρμπερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Λυπούμε ιδιαίτερος που δεν έχουμε παρούσα την Προεδρία, γιατί θέλω ιδιαίτερος να τους τιμήσω για την επιτυχία μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη αυτή αναβολή, μετάθεση της θέσης εφαρμογή. Και θέλω ιδιαίτερα ξεκινώντας ε, να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014. Λοιπόν, θα σας υπενθυμίσω, τον Απρίλιο του 2014 εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε την έγκριση της ΜΥΦΙΤΕΣ και της ΜΥΦΙΡ. Και είχαμε πει ότι περνούσαμε ένα σημείο καμπής της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είχαμε εκφράσει την υπερηφάνεια μας ε, για τον ε, Ευρωπαίο πολίτη και ψηφοφόρο που εκπροσωπούσαμε. Και λυπούμε ιδιαίτερος που δύο χρόνια μετά έρχεται η ώρα να συστήσουμε την αναβολή και να την ψηφίσουμε τώρα το μεσημέρι. Για άλλη μια φορά καθυστέρησε λοιπόν, γιατί η αρχή εποπτείας δεν ήταν σε θέση να ε, υλοποιήσει, να οργανώσει τις απαραίτητες υποδομές. Και έτσι δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε ορίσει το 2014 για την λειτουργία των νομοθετημάτων αυτών. Πρέπει να διαπιστώσουμε όμως το εξή ότι στην προηγούμενη θητεία ένα πράγμα είχαμε να κάνουμε, να φέρουμε εις πέρας, να εξασφαλίσουμε την προστασία του επενδυτή και την οργάνωση, τη σωστή οργάνωση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών μέσων. Εκεί που υπάρχει η κερδοσκοπία, εκεί που υπάρχει η ανάγκη να ρυθμιστούν οι αγορές, για να σας περιγράψω κάπως τις προκλήσεις, και μόνο από τις 3 Ιανουαρίου του 2018 βλέπουμε θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα. Λυπούμε πολύ. Από την άλλη, και πρέπει να το αναφέρω ξεκάθαρα, ότι καταφέραμε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο σε πάρα πολύ στομοχρονικό διάστημα, επί τη βάση Επιτροπής που ζητούσε την αναβολή, να εντοπίσουμε τα σημεία τα οποία είχε παραμελήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κάνουμε κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν είχαμε ξαναδεί στην Ευρώπη. Δηλαδή όλα τα προβλήματα τα οποία είχαν εντοπιστεί σε, στο επίπεδο της ε, να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι δεδομένο ότι σε κάθε κανονισμό και οδηγία που παράγει ο Ευρωπαίος νομοθέτης έχει μπορέσει να καλύψει κάθε υποπερίπτωση και ενδεχόμενο. Και πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να γίνουν μετέπειτα διορθώσεις. Εμείς από πλευράς του Κοινοβουλίου και σε αυτό θέλω ε, ρητά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες και ιδιαίτερα τους σκιώδεις συγητές με τους οποίους στενά συνεργαστήκαμε για το γεγονός ότι μπορέσαμε να εστιαστούμε, να εστιάσουμε την προσοχή μας σε εκείνα τα ζητήματα που ήταν απαραίτητο να γίνουν οι βελτιώσεις ώστε να μην ανοίξουμε ένα μπαούλο γεμάτο ζητήματα ε, και ένα τεράστιο εργοτάξιο διορθώσεων. Με το Συμβούλιο ΔΕ και την Ολλανδική Προεδρία συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και έτσι μπορέσαμε σε πάρα πολύ στομοχρονικό διάστημα να λύσουμε με εντατική εργασία πάλι τα προβλήματα που, χρήζω, που χρήζουν ε, νομοθέτησης, διορθωτικής παρέμβασης καλύτερα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί νέο νομοθέτημα. Βεβαίως πάντα υπάρχουν τέτοιες ανάγκες για βελτιώσεις και διορθώσεις και πρέπει κανείς να είναι στη θέση να παρεμβαίνει ταχύτατα σε, σε θέματα όπως αυτό. Πολλές λοιπόν οι ρυθμιστικές προδιαγραφές και πρότυπα που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό έτσι ώστε να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα το ταχύτερο δυνατό με τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Χρειαζόμαστε και θέλουμε ε, χρηματοπιστωτικές αγορές σταθερές, ε, ορθά λειτουργούσες που να αποτρέπουν τις υπερβολές και τις ακρότητες. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτόν πρέπει να τηρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Φέρμπερ, ο Χίλ έχει Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να συζητήσουμε τις τροπολογίες του MIFID 2 και αναγνωρίζω ότι έγινε πολύ σκληρή δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο για να συμφωνήσουμε από αυτόν μέχρι τον Ιούλιο. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Φέρμπερ και τους ε, σκιώδεις εισηγητές διότι διατήρησαν την όλη ορμή της προσπαθίας ε, και ήταν αποτελεσματική. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο κύριος Φέρμπερ. Αυτό το πακέτο είναι βασικό κομμάτι των ε, οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Αυξάνουμε τη διαφάνεια των αγορών και βελτιώνουμε και την εποπτεία αυτών ανταποκρίνεται στη συμφωνία των G20 στο Pittsburgh ούτω ώστε η αγορά των αξιογράφων και των παραγόγων να αναμορφωθεί, να γίνει καλύτερη αγορά, να γίνουν πιο ανθεκτικά τα προϊόντα αυτά, πιο σταθερά. Επίσης, βέβαια, θέλουμε να ενισχύσουμε και την προστασία των επενδυτών, όχι μόνο εξασφαλίζοντας το ότι οι επενδυτές έχουν τις σωστές πληροφορίες στη διάθεσή τους, αλλά εισάγοντας και αυστηρότερους κανόνες για να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων. Συμφωνούμε επί του στόχου. Και αν αυτός είναι ο στόχος, για να επιτευχθεί, χρειάζεται αυτή η νομοθεσία που πρέπει να εφαρμοστεί σωστά, με έναν τρόπο που δίδει ασφάλεια δικαίου, που δεν δημιουργεί προβλήματα για τις αγορές και επίσης προσελκύει επενδύσεις στην ευρύτερη οικονομία και μπορούν επιχειρήσεις να χειρίζονται τον κίνδυνο. Αυτή η μεταρρύθμιση πάντα θα είναι φιλόδοξη. Συλλέγει πάρα πολλά στοιχεία από πολλούς φορείς, περίπου 15 εκατομμύρια οικονομικά χρηματοστικά μέσα. Βλέποντας την κλίμακα λοιπόν του προβλήματος, τον περίπλοκο χαρακτήρα των συστημάτων πληροφορικής που απαιτούνται, θεωρείτε και σωστά ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Χρειαστήκαμε χρόνο περισσότερο για να πετύχουμε τα σωστά αποτελέσματα, όχι για να υπονομεύσουμε το νέο πλαίσιο, αλλά να λειτουργεί καλύτερα τελικά το νέο πλαίσιο όταν θα εφαρμοστεί. Το νέο αίτημα ισχύει πράγματι. Θέλουμε να παρατείνουμε την προθεσμία για την εφαρμογή του MIFID 2 κατά ένα έτος μέχρι Ιανουάριο του 2018 και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή για την υποστήριξη που μου παρήχαν και δέχονται αυτή την πρόταση που δίπεται από την κοινή λογική όπως ο κ. Φέρμπερ και εγώ είμαι ικανοποιημένο, διότι αποφύγαμε επανεξέταση των βασικών πτυχών του πακέτου που συμφωνήθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια αλλά έχουμε κάνει κάποιες τεχνικές αλλαγές στο πακέτο, αλλαγές που βελτιώνουν την ποιότητα των κανόνων, περαιτέρω διευκρίνηση του πεδίου εφαρμογή των απαιτήσεων περιδιαφωνίας για τις συναλλαγές σε πακέτα, ήταν ένα θέμα που έθεσε ΕΣΜΑ όταν υπέβαλε την έκθεσή της. Και εδώ πιστεύω ότι η τροπολογία του Κοινοβουλίου μας βοηθά να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Εξασφαλίζει ότι επικρατεί διαφάνεια πριν τη συναλλαγή, κυρίως όποτε απαιτείται, χωρίς να επιβάλλουμε ε, άχθος όταν δεν είναι κάτι τέτοιο αναγκαίο. Επίσης, σωστή ήταν η εξαίρεση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, σε αξιόγραφα SFTs από τις υποχρεώσεις για τη διαφάνεια. Τα SFTs δεν διαμορφώνουν τι τιμέ και βέβαια θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αξιόγραφα στο μέλλον. Οπότε αυξανόμενη διαφάνεια σε αυτό το τομέα θα δημιουργούσε περισσότερο άχθος χωρίς να πετυχαίνει περισσότερα πράγματα με την τροπολογία για τις εξαιρέσεις των ιδίων λογαριασμών εξασφαλίζουμε ότι οι μη χρηματοπιστωτικές εταιρείε δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του ΜΥΦΙΤ 2 χωρίς να χρειάζεται ούτε στις απαιτήσει περί και διοικητικών ρυθμίσεων εργαζόμαστε σκληρά ώστε να μπορέσουμε τα μέτρα του πέδου 2 του ΜΥΦΙΔΙΟ να τα εθετήσουμε εντός Ιουνίου. Συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Φέρμπερ ότι πράγματι θα πρέπει να διατηρηθεί ο ρυθμός αυτός. Σε διάφορους τομείς, σε κάποιους τομείς ζητήσαμε την ΕΣΜΑ να επανεξετάσει τις προτάσεις που έκανε, λαμβάνοντας υπόψη θέματα τα οποία εθίγησαν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά μαζί τα μέτρα πιστεύω ότι τελικά θα καταστήσουν το MIFID 2 αποτελεσματικότερο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σωματώσουν τα στοιχεία του MIFID 2 ε, στην ένωμη τάξη τους μέχρι τις 3 Ιουλίου του 2017 θα πρέπει ο τομέας να συμμορφωθεί από τον Ιανουάριο του 2018 ε, πιστεύω ότι είναι λογική η διαδρομή αυτή θέλουμε ομαλή εφαρμογή της νομοθεσίας και θέλουμε να επιφέρουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη προστασία των καταναλωτών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, συγγνώμη, σε αγορές στην Ευρώπη. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Χίλ. Πάμε στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Καράς, εν ονόματι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πρώτος. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Σιγητά, κυρίες και κύριοι όχι απλώς θέλουμε, απαιτείται να έχουμε, χρειαζόμαστε σταθερές χρηματοπιστωτικές αγορές. Γιατί αυτές αποτελούν την προϋπόθεση για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές που είναι απαραίτητη για να λειτουργήσουν σωστά. Οι προϋποθέσεις λοιπόν για σταθερές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι βεβαίως ρυθμίσεις κανονιστικές, διαφάνεια περισσότερη και έλεγχος. Εδώ με τη ΜΥΦΙΤ, κύριο μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έγκριση της οδηγίας ήταν η προστασία του επενδυτή. Η προστασία του επενδυτή μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν εξασφαλίζονται και οι τεχνικές προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτές τις τεχνικές προϋποθέσεις λοιπόν δεν τις είχαμε εξασφαλίσει. Είχαμε επισημάνει ότι αποτελούσε αυτό κενό, έλλειμμα και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έλεγε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτό με το σύστημα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Και έτσι το Κοινοβούλιο ουσιαστικά αξιοποίησε το χρόνο παράτασης του παιχνιδιού. Το είπε και ο κύριος Φέρμπερ και ευχαρίστησε ρητά γιατί μπορέσαμε αυτό το χρόνο της παράτασης ε, του αγώνα να τον αξιοποιήσουμε μαζί με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε να φέρουμε τις διορθώσεις. Όσο και να θέλαμε βεβαίως να ε, πούμε ότι έχουν ρυθμιστεί όλα τα προβλήματα λειτουργίας πάλι δεν είμαστε θέση να θέσουμε σε ε, λειτουργία το σύστημα και άρα για να παραμείνω στους ποδοσφαιρικούς όρους πρέπει να δώσουμε χρόνο καθυστερήσεων. Και έτσι λοιπόν πρέπει τώρα να κάνουμε μία διευκρίνηση ότι υπάρχει ο χρόνος και για την Επιτροπή και για τις επιχειρήσεις που θα χρειαστεί βεβαίως να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας τους ώστε να είναι έτοιμες μέχρι τις 3 Ιανουαρίου του 2018 να ε, εργαστούν με το νέο σύστημα. Ευχαριστώ. Κύριε Κάρας, υπάρχει μια γαλάζια κάρτα για σας. Κύριε Κάρας. There is a blue card for you. Do Θέλετε να απαντήσετε στη γαλάζια κάρτα. Κύριε Τζάνι, έχετε το λόγο. Μια ερώτηση κύριε Κάρας και ευχαριστώ πολύ που τη δέχεστε. Συμφωνούμε όλοι πως χρειαζόμαστε κανόνες διαφανείς κατανοητούς για τους πάντες, αλλά τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν η Κεντρική Τράπεζα ενός κράτους μέλους δεν τηρεί τους κανόνες αυτούς και αν δεν εισάγει σύστημα εποπτείας. Γιατί αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Η Ουγγρική Κεντρική Τράπεζα το έχει κάνει αυτό. Ο κύριος Κάρας έχει το λόγο για να απαντήσει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, οι κεντρικές τράπεζες είναι ανεξάρτητες. Και ανάλογα με την Εθνική Ένωμη Τάξη προβλέπεται έλεγχος από τα Εθνικά Κοινοβούλια και την κοινή γνώμη ασφαλώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν προκύπτουν προβλήματα μπορεί να τα συζητά ανοιχτά και στο βαθμό που το επιτρέπουν οι αρμοδιότητες τους να τα αντιμετωπίζουν. Πριν δώσω το λόγο στην κύριο Ντότς να πω ότι η συζήτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 12.30 διότι εκείνη τη στιγμή προβλέπεται να ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Παρακαλώ λοιπόν να σέβεστε το χρόνο που σας διατίθεται, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε ούτε να έχουμε γαλάζιες κάρτες, ούτε catch the eye. Συνάδελφε Ντότζ, για τους προοδευτικούς σοσιαλιστές και δημοκράτες, έχετε το λόγο. Mm. Κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, από όλα τα νομοθήματα που έχουμε θεσπίσει μετά από την χρηματοπιστωτική κρίση του 8, αυτή η οδηγία για τις κινητές αξίες και τη ρύθμιση των κεφαλαιογρών είναι η πιο σημαντική όπως είπε ο κ. Φέρμπερ. Αυτό το νομοθέτημα ή τα νομοθετήματα είναι πάρα πολύ φιλόδοξα στο τι θέλουν να καλύψουν, να φέρουν διαφάνεια στις αγορές, καλύτερη προστασία των καταναλωτών, να ρυθμίσουν κάποιες τεχνικές ε, μεγάλης συχνότητας και να σταματήσει η κερδοσκοπία σε εμπορεύματα όπως τα τρόφιμα και <clears throat> τα καύσιμα. Βέβαια θα πρέπει να δούμε το πώς μπορούμε να γυρίσουμε στα όσα ήσχαν πριν την κρίση, γιατί η κρίση αυτή ήταν τέτοια που πλήρωσαν την ύφη όλη στην Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει να δούμε για το πώς η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών θα προχωρήσει σε ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε ε, το χρονικό όριο του 2017, 30 Ιανουαρίου του 2017. Οπότε θα ήταν καλύτερο εάν το Κοινοβούλιο το συνειδητοποιήσει το πρόβλημα νωρίτερα. Ταυτόχρονα με το καινούργιο αυτό καθεστώ ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχουμε στο στόχο μα. Γι' αυτό και εγώ θα στηρίξω αυτή την πρόταση, ώστε να αναβληθεί κατά 12 μήνε η θέση σε ισχύ ε, του νέου καθεστώτο. επαναλαμβάνω δεν πρόκειται για μια πρόσκληση προ την ΕΑΚΑ προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπά στο να μην κάνουν τίποτα γιατί είπαμε ότι αυτό, το 12 μήνο είναι το ελάχιστο το οποίο χρειάζεται οπότε θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την κάθε μέρα ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η 30 πρώτου του 18 θα είναι η ημερομηνία φετηρία για την καινούργια κατάσταση. Βέβαια με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Φέρμπερ και όλους τους και όλους ήταν η συνεργασία πάρα πολύ αγαστή και έτσι μπορούμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από εδώ σε σχέση με το τι θέλουμε γιατί περιμένουμε για αυτό το δεκάμινο από Κομισιόν και ΕΚΑ. Πρώτα πρώτα αυτό που περιμένουμε είναι να έχουμε εκθέσεις πρόοδου σε τακτά διαστήματα. Να ξέρουμε ακριβώς πώς αξιοποιείται αυτό το διάστημα. Οπότε στις 30 Ιανουαρίου του 2018 ε, το μύφι, το νέο καθεστώς να μπορεί να τεθεί σε ισχύ πλήρως. Κατά δεύτερο λόγο είπαμε ότι προβληματιζόμαστε για κάποια δευτερογενή νομοθεσία επί του μύθι που θα πρέπει να δεσπιστεί και έχουμε πει τι μας προβληματίζει και αν ε, στην νομοθεσία του δευτερού επίπεδου όλα αυτά δεν λεφθούν υπόψη, τότε και εμείς θα πρέπει να κάνουμε πίσω και να απορρίψουμε. Ε, οπότε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ασχολείται και με τα παράγωγα για τα για εμπορεύματα. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα σταματήσει η χειραγώγηση των κεφαλαίων και έτσι να μην ε, φύγονται οι καταναλωτές και οι γεωργοί. Να σταματήσει η κερδοσκοπία και αυτό όσον αφορά και τις θέσεις για οποιονδήποτε παίκτη και πόσο μπορεί να κρατήσει τη θέση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα έχουμε πει επανειλημμένα. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι το όριο τήρησης της θέσης να γίνεται πιο χαμηλά και η αρχική πρόταση της ΕΚΑ δεν ήταν τόσο στεγανή, άρα σωστά την ανέπνευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλυφθούν όλα τα οποία έχει δει στο Κοινοβούλιο μέχρι ότου επιστρέψει εδώ το σχέδιο κειμένου για έγκριση ή απόρριψη. Εμείς ε, ακούσαμε και την ΕΚΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα και εκείνοι να κάνουν το ίδιο όσον αφορά αυτό το οποίο εμείς μας απασχούν για τη δευτερογενή νομοθεσία. Ο Πρόεδρος Όζογκ για την ECR. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το όνομα του ο στόχος είναι να βληθεί θέση σε ισχύ της οδηγίας το 2014 κατά ένα δωδεκάμινο συνολικά. Τελικά θα τεθεί σε ισχύ το 2018. Είναι περιπλοκότατο το θέμα και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν είναι εξίσου περίπλοκα. Υπάρχει και ανάγκη για τεχνικές υποδομές Επίσης, οι διάφοροι φορείς σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και εκτός αυτού χρειάζονται το 12 αυτό. Η εφαρμογή και η υλοποίηση της υποδομής θα περάσει από πέντε φάσεις. Μεταξύ αυτών των φάσεων έχουμε και τις διάφορες δοκιμές και την όλη διαμόρφωση των προγραμμάτων. Μέχρι τον Ιούλιο φέτος χρειαζόμαστε να τα ετοιμάσουμε όλα, θέλουμε να τα δοκιμάσουμε και να λειτουργούν όλα σωστά. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούν σωστά. Εν ονόματι τώρα τη ομάδα των φιλελευθέρων, συνάδελφε Βαν αν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω τον Μάρκους Φέρμπερ, τον εισηγητή Η συνεργασία μαζί του είναι πάρα πολύ δημιουργική. Αποτελέσαμε μια ομάδα διαπραγματεύση κατά αυτή την ε, δύσκολη περίοδο για αυτές τις ακαθόδες συζητήσεις ε, είχαμε έρθει σε επαφή και με τις αγορές αλλά και με κροσούς καταναλωτών και των εταιριών που εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε ήταν δύσκολο να μπορέσουμε να πετύχουμε μια εξισορρόπηση συμφερόντων. Και βέβαια η Ένωση κεφαλαίων ε, ήταν πάρα πολύ, ε, είχε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο και οπότε θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν τόσο ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ο κύριος Τίμερμανς στο θεματολογιό του ήθελε καλύτερη νομοθεσία. Βέβαια όσον αφορά τώρα το MIFID ε, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα πώς θα πετυχούν το στόχο μας και για το MIFID ισχύει το ίδιο και θέλουμε να είναι ενημερωμένοι καταναλωτέ όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τι κινητέ αξίε, τι επενδύσει του τέλο πάντων, ούτω ώστε να μπορούν ε, με τα λόγω γνώσεω να λάβουν τι αποφάσει του. Και επίση δώσαμε πραγματικό αγώνα, πραγματική μάχη ή γι' αυτό και καθυστερήσαμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Βέβαια, είναι κατανοητό το γιατί έγινε αυτό, γιατί θέλουμε κάποια ρύθμιση που να μην είναι, να είναι κάποια ρύθμιση η οποία να αποδίδει. Να, γιατί υπήρξε η καθυστέρηση, να γιατί τώρα έχει ζητηθεί αυτή η αναβολή και όπως είπε και η κυρία Ντότζ, θα πρέπει να καταλήξουν σε κάτι το οποίο να λειτουργεί εύρευμα σαν ρύθμιση. Λέμε τώρα για έρευνα. Τι είπα να πει έρευνα. Δεν είναι κάτι το έλασο, είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτό το νομοθέτημα. Άρα χρειάζεται ξεκάθαρη ρύθμιση, ξεκάθαρος ορισμός του τι είναι έρευνα. Θα πρέπει ο κόσμος να έχει ενημέρωση όσο γίνεται πιο επικαιροποιημένη. και για κάποιες ε, συναλλαγές που έχουν πραγματικά λάβει χώρα και έτσι να λαμβάνονται οι αποφάσεις για επενδύσεις. Όπως είπε ο βέβαια όλα τα πολύτιμα πράγματα δεν επιδέχονται όλα υπολογισμό και αποτίμηση, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι το ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους φορείς των καταναλωτών, της προστασίας καταναλωτών και τελικά να καταλήξουμε σε λύση ευμενή για τους καταναλωτές και τους επενδυτές. Επίσης αυτός ο κλάδος να μην ε, εμποδίζεται από προβλητική γραφειοκρατία. Και τώρα για την ΚΟΕ. Ο κύριος Ντεμάζη. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Μια δεκαετία μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης ακόμα δεν έχουν θεσπιστεί τα απαραίτητα νομοθετήματα. Με βαριά καρδιά η ομάδα μου υποστήριξε την αναβολή της θέση εφαρμογή, ε, εφαρμογής γιατί βλέπουμε ότι και πάλι τα χρηματοπιστωτικά λόμπι πέρασαν τη δική τους γραμμή. Η ΑΚΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη δεν έχουν προσαρμόσει τον τρόπο δράσης τους στα τελευταία ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Και επιπλέον το σύνολο του χρηματοπιστωτικού όγκου δεν ελέγχεται, δεν ελέγχονται κινήσεις μέσω των ΗΠΑ και δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ισότιμη ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βάζουμε τους σπόρους για την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμπέρτς έχει το λόγο. Μέρος των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Έχουν περάσει 9 χρόνια μετά την αρχή της ε, χρηματοστοιχική κρίση σήμερα. Ονομαστικό όγκο των χρηματοστοιχικών αγορών καθημερινά είναι 10 φορέ το μέγεθος της πραγματικής οικονομίας, δεκαπλάσιος. Υπάρχει 10 φορέ περισσότερη κερδοσκοπία για ένα δολάριο του εμπορίου. Για κάθε δολάριο κερδοσκοπία είναι 10 δολάρια. Αυτές οι δραστηριότητε είναι άχρηστες και παρενοχλούν την πραγματική οικονομία, κυρίως όπως είπε η κυρία Ντότζ Καθημερινά γίνεται κερδοσκοπία επί των πρώτων υλών και κυρίως των τροφίμων, των πρώτων υλών των τροφίμων. Είναι απίστευτο αυτό που διαπιστώνουμε. Ένα κείμενο που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 για να εφαρμοστεί αρχές του 2017, δηλαδή τρία χρόνια αργότερα, ακόμα να είναι έτοιμο να εφαρμοστεί σε ένα εξάμεινο. Και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 18 μήνες με την θέτηση του εγγράφου ε, ζητά την αναβολή ε, για ένα χρόνο. Αυτό δείχνει την, τον υπερβολικά περίπλοκο χαρακτήρα του κειμένου και τη χαλαρότητα. Μια απλή νομοθεσία και πιο αυστηρή θα ήταν καλύτερη από μια υπερβολικά περίπλοκη νομοθεσία και λόγω της περιπλοκότητας μας ζητάνε έναν χρόνο παραπάνω. Και σαν να μην και αν ήταν μόνο αυτό θα λέγαμε έστω. Δεν ήταν πολλοί επαγγελματίε στην ε, προσέγγιση τους. Ας τους δώσουμε ένα χρόνο. Αλλά ένας χρόνος παραπάνω είναι ένας χρόνος παραπάνω ε, κερδοσκοπίας. Κυρίως όσον αφορά τα τρόφιμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή, αυτό το κείμενο ήταν ευκαιρία να περάσουν νέε εξαιρέσει που θα μειώσουν περισσότερο τη διαφάνεια των χρηματοδοτικών αγορών. Όλο τυχαίω. Διαθετώντας αυτές τις εξαιρέσεις, επιβεβαιώνουμε την υπόνοια ότι αυτές οι καθυστερήσεις χρησιμοποιούνται για να αποδυναμωθεί ένα κείμενο που πάλι δεν ανταποκρινόταν στις φιλοδοξίες μας. Εμείς θα καταψηφίσουμε συνεπώς αυτή την καθυστέρηση, αν υπήρχε μόνο αυτή, διστακτικά θα υπερψηφίζαμε. Αλλά εδώ, λόγω των συμπληρωματικών εξαιρέσεων που ε, υποβάλλει το κείμενο αυτό, αρνούμεθα να το υπερψηφίσουμε, τα απορρίπτουμε. Ευχαριστώ. και Συνάδελφε Βάλλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι είναι περίπλοκο το να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις αιμοτοπιστωτικές αγορές, αλλά όλο αυτό τον χρόνο που διαθέσαμε για να το καταφέρουμε είναι χρόνο που δεν τον έχει ο κόσμος όπως ο κ. Λάμπερτς και ακριβώς η αγορά ε, λόγω της ε, κρίσης τώρα έχει φουσκώσει. Ε, ξεκίνησε αυτή η διαδρομή το 2008-2009 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να δώσει μια όθηση στην κεφάλαια αγορά και θεώρησε ότι τα μέτρα για τις τράπεζες, για την πραγματική οικονομία έχουν θέματα προτεραιότητας και αυτό αποδεικνύει ότι στην σημερινή Ευρώπη του Ιούνκερ ε, η Ευρώπη τελικά εκπροσωπεί τα δικαιώματα των ισχυρών, των ε, τραπεζών και όχι των Ευρωπαίων πολίτων. Να, και τώρα λοιπόν έχουμε την πρόταση παράταση της θέση σε ισχύ. Ε, αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά και από την άλλη μεριά πρέπει να εκμεταλλευτούμε εδώ το χρόνο να κάνουμε κάποιες ε, τροποποίησεις όπως είπαν οι συνάδελφοι από τους πράσινους αλλά αυτό θα να μην είναι μόνο της ε, τράπεζας. χρειάζεται κάποια διαφάνεια και όσον αφορά τους χρηματομεσίδες και να ρυθμίσουμε και τα παράγωγα για κάθε ε, χρηματοπιστωτική συναλλαγή και όλα αυτά που σημαίνουν κάποιες προμήθειες για τις τράπεζες, όλα αυτά να διέπονται από διαφάνεια. Όλα αυτά είναι συστημικού χαρακτήρα και θα πρέπει όλα αυτά να μην κοστίζουν στους φορολογούμενους και ξέρετε ότι εδώ θέλουμε διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές. Οπότε αυτό το οποίο εμεί θέλουμε είναι να είμαστε αποφασιστικοί όσον αφορά τα μέτρα για τις τράπεζες και όσον αφορά τις ρυθμίσεις σχετικές με τις συναλλαγές. Ακριβώς όπως ελέγχθη, πρόκειται για κάτι πολύ δύσκολο. Ευρώπη των Εθνών και των Ελευθεριών, κυρία Κάπελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επίτροπε Χίλ. Συμφωνούμε σήμερα ότι η μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, δηλαδή η ρύθμιση χρηματοπιστωτικών μέσων πρέπει να αναβληθεί κατά ένα χρόνο και όντως πρέπει και γι' αυτό ε, θα συμφωνήσω. Ωστόσο θα συμφωνήσω και με τις επικρίσεις του ε, εισηγητή ότι δεν μπορούμε να δώσουμε κανένα άλλο περιθώριο καθυστέρηση στην Επιτροπή και την ΑΚΑ. Ο χρηματοπιστωτικός χώρος πρέπει να είναι ε, έτοιμος για να προσαρμοστεί στους όρους της MIFID, του MIFID, του κανονισμού MIFID, για να μην υπάρξουν νέα προβλήματα, για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη διαφάνεια. Διαφάνεια, προστασία των επενδυτών και εδώ ακριβώς χρειάζεται να καταγράφονται οι εκθέσεις των τραπεζών για τις δραστηριότητες τους και των λοιπόν βεβαίως ε, ιδρυμάτων και πρέπει να ε, εξασφαλίζεται η λειτουργία τους με ίδια κεφάλαια. Τα, τα, οι όγκοι των συναλλαγών επίσης πρέπει να είναι δυνατόν να παρακολουθηθούν. Πρέπει να υπάρχουν όρια θέσεων ανάλογα με το προϊόν, ιδιαίτερα στην διαπραγμάτευση πρώτων υλών, που όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν είναι χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν μπορούμε, όπως είπε και ο Επίτροπος, να μιλούμε για χρηματοπιστωτική διαπραγμάτευση των ε, πρώτων υλών κατά αυτούς τους όρους. Ο κύριος Φουντούλης έχει το λόγο. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει πως, όπως πάρα πολλοί τομείς της οικονομίας, έτσι και η αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων έχει ανάγκη συγκεκριμένων ρυθμίσεων, ώστε να καταστεί ασφαλέστερη για όλους όσους επιλέγουν να δραστηριοποιούνται σε αυτήν αρχικά για τα κράτη μέλη της ένωσης και την αποφυγή τελέσεως παράνομων πράξεων και εν τέλει για το καλό των κοινωνιών μας στο σύνολό τους. όμως όσο αναγκαίες και αν είναι κάποιες από τις ρυθμίσεις αυτές όσο και αν έχουν προβλεφθεί τυχόν κενά η αλήθεια είναι πω σε τίποτα δεν θα επηρεαστεί προ το καλύτερο η καθημερινότητα του απλού πολίτη. η ανεργία αυξάνεται και η φτώχεια χτυπάει την πόρτα κάθε μέρα σε περισσότερε οικογένειε δυστυχώ εν μέσω τη κρίση που διέρχεται τα τελευταία δέκα χρόνια η ευρώπη οι πολίτε απαιτούν δραστικέ λύσει στα καθημερινά του προβλήματα. εκθέσει όμω όπω αυτέ για τι οποίε συζητάμε σήμερα δεν προσφέρουν τι λύσει αυτέ. θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση των πολλών σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων των ευρωπαίων πολιτών πέρα από τι στοχευμένε παρεμβάσει στόχος της έκθεσης είναι να ενισχύσει την προστασία των επενδυτών με τη θέσπιση ισχυρών οργανωτικών απαιτήσεων και απαιτήσεων συμπεριφοράς θέματα όμως μικρής σημασίας για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. ο λόγος για τον οποίο οι πολίτες της ευρώπης μας επέλεξαν για να τους εκπροσωπούμε εδώ είναι να δίνουμε λύση στα καθημερινά τους προβλήματα και περιμένουν αποτελέσματα τα οποία δυστυχώς το σώμα αυτό δυσκολεύεται πάρα πολύ να παρουσιάσει μιας και είναι ελάχιστα τα όσα έχετε καταφέρει να κάνετε πράξη προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων μέχρι σήμερα. ευχαριστώ. Ο κύριος Κίρτσος το λόγο. κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι αναγκαία η παράταση την οποία θα ψηφίσουμε οι περισσότεροι από εμά. Ταυτόχρονα όμως τη θεωρώ μία ήττα θα μπορούσαμε να πούμε των ευρωπαϊκών θεσμών με την έννοια ότι δεν παρακολουθούμε μία πραγματικότητα με τους ρυθμούς που αυτή εξελίσσεται. Έχουμε μία θεσμική βραδύτητα στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων είχαμε τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, την οποία πλήρωσε ιδιαίτερα ακριβά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε μέσα από τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες που είχε την ίδια τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κινδυνεύουμε λοιπόν να παρέμβουμε το 2018 χωρίς να υπάρχει καμία εγγύηση ότι μέχρι τότε δεν θα υπάρξει μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση αρκεί να δούμε τι γίνεται για παράδειγμα στην κίνα αρκεί να δούμε τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος στον ευρωπαϊκό νότο αρκεί να δούμε τις δυσκολίες που έχουν οι τράπεζες με τα αρνητικά επιτόκια τις δυσκολίες των ασφαλιστικών εταιριών ε, ακόμα και τις δυσκολίες που θα προκύψουν στις ηνωμένε πολιτείες και στο ηνωμένο βασίλειο δύο πανίσχυρα χρηματοπιστωτικά κέντρα εξαιτία των ε, πολιτικών εξελίξεων. επομένω κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε μια μεταβατική άμυνα δηλαδή πώ θα πάμε από τη μία περίοδο στην άλλη του αυστηρότερου ελέγχου χωρί να πάθουμε μεγάλη ζημιά. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, συνάδελφε Γκραπίνη. Δεν μπορούσα να δώσω γαλάζια κάρτα. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Έχουμε καθυστερήσει 12.30. Πρέπει να ψηφίσουμε, βλέπετε και αν τα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τι 12.30. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να επιτρέψω γαλάζιες κάρτες. Συνάδελφε Γκουαλτιέρη, έχετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σημερινή ψηφορία ολοκληρώνει με επιτυχία μια διαδικασία κρισίμου σημασία για την ολοκλήρωση τη ρυθμίσεω για τι χρηματοστατικέ αγορέ Ευρωπαϊκή Ενώσεω. ΜΥΦΙΡ και το ΜΥΦΙΡ είναι πυλώνε βασικοί αυτού το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πέτυχαν μια σημαντική συμφωνία που εγγυάται τη σταθερότητα και τη βεβαιότητα στους φορείς της αγοράς και τις εποπτικές αρχές και τα κράτη-μέλη δεχόμενη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καθυστερήσει για μια χρονιά η εφαρμογή αυτού του νομοθετικού πακέτου και ενσωμάτωση οδηγία στην ένωμη τάξη των κρατών μελών στις διάφορες αρχές να δημιουργήσουν τις κατάλληλε υποδομές και το λογισμικό για να συλλεχθούν τα κατάλληλα στοιχεία για την εφαρμογή των νέων μέτρων. Το Κοινοβούλιο ήταν συνεκτικό διότι ολοκλήρωσε γρήγορα ε, και με αποτελεσματικό τρόπο την διαδικασία χάρη στην πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου και των εισηγητών υποστηρίζοντα τη διαπραγματευτική ομάδα αυτή η ταχεία διαδικασία επέτρεψε να γίνουν και σωστέ τροπολογίε στο κείμενο και έτσι η εφαρμογή θα είναι πιο συνεκτική και θα πετύχουμε του στόχου ε, τη νομοθεσία μαζί με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτή η πρόταση θα, ε, θα καλούσα τον κύριο Λάμπες να διαβάσει περισσότερο τα κείμενα σχετικά με αυτό και να μην είναι αντιπαραγωγικός λέγοντας πράγματα που δεν είναι σωστά. Αν δει ποια είναι η φύση των αλλαγών που έγιναν που πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή γίνεται πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό το κείμενο του νομοθετήματος. Υπογραμμίζω εξάλλου ότι για για την καλύπτεται από τον κανονισμό για τις σηματοστικές συναλλαγές η ανταλλαγή αξιογράφων ε, και δεν χρειάζεται να καθορίζονται τιμές. Το MIFID είναι βασική σημασία για την προσπάθεια εναρμόνιση τη αρχιτεκτονικής αρχιτεκτονική τη Ενώσεω και για τη δημιουργία του ενίου ε, οδηγού rule book που είναι απαραίτητο για να υπάρχει μια ενιαία ε, αγορά επενδυτικών υπηρεσιών και για τις κεφαλαγορές. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάγκη τάχιστα να υιοθετηθεί η νομοθεσία σε δεύτερο επίπεδο που είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εγγυάται την πλήρη εφαρμογή όλων των μέτρων από την 1η Πρώτου του 2018. Συνάδελφε Μέσο Σμιτ. Η σημερινή πρόταση νόμου είναι μια παρέμβαση αναγκαία όσον αφορά τις ε, αγορές των επενδύσεων. Γι' αυτό και εμείς θα την επιψηφίσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα οριοθετήσουμε τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, διότι έχουν οδηγήσει ε, σε πάρα πολλές διαταραχές στις ε, αγορές. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις συναλλαγές για τα παράγωγα εμπορευμάτων που έχουν σχέση με τη διατροφή, επίσης με τις ε, πρώτες ε, ύλες. Αυτό στην αρχή νομίζαμε ότι θα ωφελήσει τους Γιώργου οδήγησε όμως σε μια φούσκα σε μια τιμολογική πολιτική που ξέφυγε και ήταν τραγικές οι συνέπειες άρα είναι καλό πάλι καλά τέλος πάντων καλό, καλή αργά παρά ποτέ που τώρα έχουμε μια ρύθμιση που θα οδηγήσει σε χρηματοπιστωτικές αγορές που θα είναι πιο δίκαιες και θα λειτουργεί καλύτερα το σύστημα και τώρα κύριε Ματίας έχει το λόγο λέει ο Πρόεδρος Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια από την ε, κρίση άρα ήρθε η ώρα να σταματήσουμε απλώς να χρυσώνουμε το χάπι και η συζήτηση που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι βέβαια δικαιολογημένη, όμως τίποτα δεν άλλαξε. Τελευταία δέκα χρόνια τίποτα δεν άλλαξε. Έχουμε 50 εκατομμύρια ε, διαφορετικά είδη κινητών αξιών και θα πρέπει να δούμε το πώς θα σταματήσουν πλέον την ύφη οι πολίτες για την κρίση αυτή, γιατί δεν φταίνε εκείνοι. Έχουμε ένα σωρό επομένω ε, μέσα πολιτικής, εξαιρέσεις, παρεκκλήσεις. Ε, υπάρξει και κάποια στεγανή νομοθεσία τελικά. Τελικά η δημοκρατία μας έχει πέσει όμοιρος των χρηματοοικονομικών ομίλων. Χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη ρύθμιση. Η οδηγία MIFID θέλει να εμποδίζει τι τράπεζε να πουλήσουν οτιδήποτε σε οποιονδήποτε, δηλαδή ε, αξιόγραφα με υψηλό κίνδυνο σε κίνδυνο σε πελάτε που είναι ευάλωτοι και είναι καλά πληροφορωμένοι. Η έκθεση που θα ψηφίσουμε θέλει να αναβάλει την εφαρμογή τη οδηγία για το 2018, δηλαδή 10 χρόνια μετά την κρίση των subprimes. Και θέλουμε να δώσουμε και άλλη καθυστέρηση για τι τράπεζε που καταχρώνται την αξιοπιστία των ιδιωτών και των επιχειρήσεων που είναι καμιά φορά έφραυστη. Ή το ένα ή εφραστη. η Ευρωπαϊκή Ή η ευρωπαικη αρχη των Αγορών, πλάσμα δεν είναι αρμόδια για να θεσπίζει σοβαρή νομοθεσία για την είτε δίνει στι μεγάλε πολυεθνικέ τράπεζε περαιτέρω ανάσα για να συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται διάφορα κενά τη παρούση νομοθεσία. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον τομέα όπω και σε άλλου, δεν θα έπρεπε να δίνουμε υποσχέσει που δεν να τηρηθούν, διότι στο ανέφικτο τίποτα δεν επιτυγχάνεται. Πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταπολεμήσει την απακτικότητα των τραπεζών, ενώ ε, κάνουν ελεύθερε συναλλαγέ ανεξέλεγκτα. Πέρα από τις δηλώσεις επί της αρχής, το δική σας υποφιλελεύθερο λογισμικό σας δεν σας επιτρέπει να πλαισιώσετε καλύτερα τις διάφορες δραστηριότητε που είναι κυρίως κερδοσκοπικές. Συνάδελφε Τόμκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λυπούμε που δεν μπορεί να υλοποιηθεί το 2017 όπως είχε προβλεφθεί αρχικά η οδηγία. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την προστασία του επενδυτή πρέπει να δώσουμε αυτήν την εγγύηση, αυτήν την παράταση. Ε, η χρηματοπιστωτική κρίση μας έχει διδάξει πολλά. Έχουμε εντοπίσει στο χρηματοπιστωτικό ρυθμιστικό πλαίσιο πολλά σημεία κενού, αδυναμίας, που πρέπει να καλυφθούν ώστε να καταπολεμηθούν οι μη σοβαρές πρακτικές, ώστε να προστατευτεί καλύτερα ο επενδυτής. Χρειαζόμαστε καλύτερες δομές επενδυτικές, εμπορικές, περισσότερο έλεγχο και αρμοδιότητες για την εποπτεία των αγορών. Όλα αυτά για να προστατευθεί καλύτερα ο καταναλωτής, ο επενδυτής. και ένα σύστημα δεδομένων, συλλογής δεδομένων, που θα μας εξασφαλίσει περισσότερη διαφάνεια επίσης. Και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτούς τους λόγους που εξέθεσα υποστηρίζω τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Τζιλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Σιγητά, είναι σημαντικό το ότι μπόρεσε το Συμβούλιο μαζί με το Κοινοβούλιο να εξεύρουν μια συμβαστική λύση για την υπόθεση αυτή. Το MIFID, και το MIFID, είναι, το MIFID 2 και το MIFID είναι τα δύο μεγάλα νομοθετήματα για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες και να προβλεφθούν και να αποτρεπούν στο μέλλον ε, χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Αυτό σημαίνει εισαγωγή νέων κανόνων εδώ. Ωστόσο, λυπούμαστε γιατί θέματα υποδομών πληροφορικής ουσιαστικά δεν μας επιτρέπουν να θέσουμε σε εφαρμογή και μας εξαναγκάζουν να αναβάλουμε για ένα χρόνο τη ΜΥΦΙΤ 2 και τη ΜΥΦΙΡ. Μας λέει η Επιτροπή λοιπόν ότι ε, θα είναι έτοιμη σε ένα, χρόνο, σε ένα μισό χρόνο από τώρα, από τον Ιανουάριο του 2018. Μακάρι, μακάρι, γιατί πραγματικά θα αισθανθούμε μεγάλη απογοήτευση εάν δεν είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία όλη αυτή η νομοθεσία στον Ιανουάριο του 2018. Δεν πρέπει να δοθεί άλλη αναβολή. Μέτρα λοιπόν που θα καταγράφουν, που θα ε, λαμβάνουν υπόψη τα μελήματα του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα για το νέο καθεστώς το σχετικό με τα παράγωγα και τις αγορές βασικών αγαθών που θέλουμε να μην επηρεάζουν την τιμή στον καταναλωτή. Και αυτό όχι μόνο για τους ψηφοφόρους της δικής μου περιφέρειας, αλλά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης θέλουμε η Επιτροπή να προσδιορίσει σε λεπτομέρειες το νέο καθεστώς σε επίπεδο 2 και όχι να υποβαθμίσει σε επίπεδο ε, πρώτο τις φιλοδοξίες όπως τις έχουμε εμείς περιγράψει. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας Επίτροπε. Μα ζητάτε λοιπόν να αναβληθεί αυτό το πακέτο έως τις 3 ε, Ιανουαρίου του 2018 για να γίνει σωστά η δουλειά, για να ρυθμιστούν τα πάντα. Καλύτερα αυτό βέβαια από το να γίνουν ταχύτερα και με ανεπαρκή τρόπο εδώ έχουμε να κάνουμε με τις συνέπειες της μεγάλης ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ύφεσης που ακολούθησε. Προφανώς θέλουμε μια ορθώς λειτουργούσα χρηματοπιστωτική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι απαραίτητη για τις αγορές μας, για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο αυτές οι αγορές χρηματοπιστωτικές πρέπει να λειτουργούν σωστά με βάση τους κανόνες. Ιδάλλως μπορεί να καταστρέψουν την οικονομία. Χρειάζεται περιβάλλον προστασίας του καταναλωτή, του επενδυτή. Χρειάζεται περιβάλλον διαφάνειας. Όλα αυτά χρειάζεται να γίνουν και έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και καιρό πολύ. Έχουμε καθυστερήσει. Χρειάζεται ένα σύστημα ενημέρωσης, αποκάλυψης και καταγγελίας των ε, κακόπιστων και κακοπροαίρετων ε, πρακτικών, τη παράβαση των κανόνων. Πρέπει να προστατεύεται ο καταναλωτή και ο επενδυτή από εκείνον που κερδοσκοπεί εις βάρος του. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση των οικονομιών μα αυτή η νομοθεσία. Να μας, θα μα επιτρέψει να αποφύγουμε τι κερδοσκοπικέ φούσκε που θα μα ρίχνουν και πάλι στην ε, ύφεση. Σα ευχαριστώ πολύ και υποστηρίζω τι τροπολογίε. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Συνάδελφε Σαντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κείμενο που συζητούμε αφορά περίπλοκους κανονισμούς που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στον απάντηση στις απαιτήσεις της χρηματοστηρικής αγοράς στην Ευρώπη και αλλού. Έχουμε έτσι τη δυνατότητα να σκεφτούμε τον τομέα αυτών, τον χρηματοστηρικό με τον οποίο σχετίζονται τα μέτρα τα πρόσφατα χρόνια, κυρίως μετά τα Lux και τα σκάνδαλα του Panama Papers, τα χρηματοδοτικέ υπηρεσίε, στα μάτια των απλών ανθρώπων σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, ξέπλυμα χρήματο και διαφθορά. Θεωρούνται ότι το χρησιμοποιούν ε, αδίσταχτοι τραπεζίτε και λογιστέ που θέλουν να προωθήσουν του φορολογικού παραδείσου και να έχουν κέρδη. Αυτή είναι μια εντύπωση, αλλά απέχει από την πλήρη αλήθεια. Το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε και η Ευρώπη που δημιουργείται χρειάζονται χρηματοδοτικέ υπηρεσίες που είναι ακέραιες, ούτω ώστε οι διαθέσιμοι να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Αυτό δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Εδώ δημιουργούμε νέε μεθόδου που καθιστούν χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε προσαρμοσμένε στι σημερινέ και ανάγκε. Όμω χρειαζόμαστε νέα μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι βέλτιστε πρακτικέ χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε καθορίζονται από επαγγελματική συμπεριφορά που θέλει να χρησιμοποιείται σωστά δεντολογικά. Μέχρι του παρόντο δεν είχαμε τέτοιε διαβεβαιώσει. Συνάδελφε Κοτσολίνο, έχετε το λόγο εδώ που βρίσκουμε δεν μπορούμε να πετύχουμε του 2018 για να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Θέλουμε αποτελεσματικότερη συλλογή στοιχείων και για την αρμόδια αρχή συνοδευτική υπηρεσία και για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είμαστε πιο συνετοί όμω αφορά την προσέγγιση. Όταν θεσπίζουμε μεταρρυθμίσει αυτή τη εμβελία χωρί να καθορίζουμε στόχου χρονικού αξιόπιστου και σίγουρου χωρίς να θετούμε μέτρα επαρκή που θα εγγυούνται τη μεταβατική φάση. Παραδείγματο χάρη, θα δώσουν δυνατότητα στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Αρχή να έχει ανθρώπινου πόρου και οικονομικού. Έτσι βοηθούμε του κερδοσκόπου. Θέλουμε να βοηθήσουμε του καταναλωτέ και του ομοταμιευτέ. Θέλουμε να κάνουν πιο αξιόπιστη την μάχη για τι ε, ε, χρηματιστικέ αγορέ που να γίνουν πιο διαφανεί. Δεν μπορούμε να έχουμε φιλόδοξου στόχου στην νομοθεσία και να εγκαταλείπουμε τελικά την νομοθεσία. Η αναβολή για ένα χρόνο λοιπόν δεν είναι μια υποχώρηση, είναι μια αναγκαιότης που δεν θα την σπαταλήσουν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς και θεσμοί. Συνάδελφε Μορέλ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, βέβαια και η ρύθμιση των αγορών ήταν κάτι επιτακτικής σημασίας, κάτι που αφορά σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους, όλους οι οποίοι έγιναν μάρτυρες και θύματα όλων αυτών των διαδοχικών κρίσεων από το 8 και είδατε ε, το πόσο κυρίαρχη θέση απέκτησαν κάποια, ε, κάποιες κινητές αξίες, τόσο κάποια μέσα συναλλαγών σε χρηματιστήρια. Άρα δεν θέλουμε με τίποτα να δώσουμε επιταγή λευκό στην Επιτροπή και να αναβάλει και να εγκαταλείψει τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων και κατά νου. Έχω ε, το τι γίνεται από κερδοσκοπία με τις συναλλαγές για τα τρόφιμα. Τέλος, δεν είναι δυνατόν να κλείνω μία πόρτα για να ανοίξει περισσότερο άλλη ε, και εμείς ως σοσιαλδημοκράτες δεν θέλουμε να υπάρχει τιτλοποίηση και η οποία να γίνεται ε, με τυφλό ε, τρόπο όσον αφορά τις κεφαλαγορές. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Πάντως γενικά το κείμενο έχει την σωστή ρότα. Κάτσε διάρκεια, τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προστασία του καταναλωτή, προστασία του επενδυτή του πολίτη, ανάκτηση της ε, εμπιστοσύνης, καταπολέμηση της ε, κερδοσκοπίας, διαφάνεια στις ε, συναλλαγές. Όλα αυτά είναι το θεματολόγιο, η στόχη μας. Η κρίση του 8 αφορούσε τα ρίσκα ενός αχαλήνα του συστήματος που τελικά έθιξε την πραγματική οικονομία κυκλοφορούν ε, χρήματα που δεν είναι πραγματικά, ε, αλλά με την ταχύτητα του φωτό γίνονται αυτέ τι συναλλαγέ. Αυτό επομένω ας σταματήσει ε, και θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματική νομοθεσία κατά της κερδοσκοπίας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Οπότε εδώ μας ζητούν ότι θα πρέπει με αυτή την παράταση να ρυθμίσουμε κάποιες λεπτομέρειες και να ελπίσουμε στο μεταξύ θα έχουμε νέα κρίση. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Η τιμολόγηση των χρηματοδοτικών μέσων και συμβολέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο ακριβή θα είναι τα στοιχεία αναφοράς. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία αναφοράς σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και για τον λόγο αυτό η ευρωπαϊκή αρχή κινητών αξιών και αγορών και οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα δεδομένων αναφοράς χρηματοδοτικών μέσων ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων. φυσικά οι αρμόδιες αρχές θα λειτουργούν υπό την κατάλληλη εποπτεία ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια ορθή όρη τιμολόγησης και εξάλληψη φυσικά οποιασδήποτε περίπτωσης κατάχρησης της αγοράς. άλλωστε η επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει απαιτήσει που αφορούν την αδειοδότηση και την λειτουργία των επιχειρήσεων παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και αναφορά δεδομένων. όμω δεδομένου ότι οι υποδομέ συλλογή των απαραίτητων αυτών στοιχείων δεν είναι έτοιμε μέχρι τι προβλεπόμενε ημερομηνίε ο κανονισμό που προτείνει η επιτροπή μπορεί να μεταφερθεί ένα έτο αργότερα ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε του συστήματο οι συνδιαλλαγές στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων λόγω της φύσης τους περιέχουν μεγάλο επιθετικό ρίσκο. η ανέδεια δεν αποτελεί δικαιολογία είναι όμως τεράστιο ηθικό αμάρτημα αν θέλετε ποινικό αδίκημα όταν αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης ανθρώπων που απλά αναζητούν ευκαιρίες επένδυσης. οι επιχειρήσεις παροχής επιθετικών υπηρεσιών οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων λειτουργούν με ιδιότυπους κανόνες και εκτός πλαισίου οποιασδήποτε εναρμονισμένης πρακτικής. συχνά λειτουργούν ως δεκανίκη μεγάλων τραπεζικών κολοσσών αλλά και κυβερνήσεων με σκοπό να συλλέξουν χρήματα πολιτών οι οποίοι δεν είναι καταθέτε. Τρανό θυμήθηκε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όταν χιλιάδε πολίτε παρασυρώμενοι από ένα κλίμα εφορία που εντέχνω δημιούργησε τότε η κυβέρνηση με ψέματα και φρούδε ελπίδε, επένδυσαν του κόπου του σε εταιρείε φαντάσματα και μετοχέ φούσκε. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών οφείλει πρωτίστω να επιβάλλει του κανόνε διαφάνεια και του βέλτιστου κανόνε εκτέλεση των συναλλαγών. Κυριότερα όμω πρέπει να θεσπίσει ένα πλαίσιο κυρώσεων σε αυτούς που χρησιμοποιούν αθέμητα μέσα ακόμα και παραπληροφόρηση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στις αγορές και να χάνουν χρήματα οι ιδιώτες επενδυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από το βασικό στοιχείο που αναφέρθηκε για τις αρχές, για τις καλές ρυθμίσεις. Δηλαδή θέλουμε να καθορίσουμε ρεαλιστικές προθεσμίες και να τις πετύχουμε. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω τις προθεσμίες. Άκουσα ξεκάθαρα τις εκφραστήσεις απόψεις. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που μου δώσατε σε αυτή τη φάση όπου ακολουθήσαμε την κοινή λογική. Δηλαδή ότι χρειάζεται η καθυστέρηση ούτω ώστε αυτό το περιπλοκότατο νομοθέτημα να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί σωστά. Αυτή είναι η σωστή απόφαση. Αλλά είμαι, σας υπόσχομαι ότι θα τηρήσουμε τις προθεσμίες που θέσαμε. Θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές οι προθεσμίες ε, για να εφαρμοστούν τα μέτρα γέρος. Όσον αφορά τις διάφορες λεπτομέρειες, προσπαθούμε τα περισσότερα μέτρα του επίπεδου 2 να τον Ιούνιο Ήδη υιοθετήσαμε 11 μέτρα και τα υπόλοιπα θα υιοθετηθούν αυτό το μήνα. Πράγματι ζητήσαμε σε κάποιους τομείς η αρμόδια Ευρωπαϊκή Αρχή να εξετάσει τις προτάσεις και αυτό αντικατοπτρίζει θέματα που έχουν τεθεί από το Κοινοβούλιο. Επανεξετάζουμε κάποιες απαιτήσεις περί διαφανείας για ομόλογα και αγορές παραγόγων. Ζητήσατε πιο συνετή προσέγγιση, κατά την άποψή μας αυτό το εγγυόμεθα και ζητείτε και για τις, ε, διάφορα, τα διάφορα όρια ε, που ανέφεραν διάφορα μέλη. Για τα γεωργικά παράγωγα θέλουμε οι θέσεις, τα όρια για τις θέσεις να είναι πιο ευαίσθητα και για τις πολύ μεταβλητές αγορές και για τις λιγότερο ευμεταβλητές. Κάποιοι στο Κοινοβούλιο θέλουν να περιοριστήσει η υπερβολική μεταβλητότητα και κερδοσκοπία στα διάφορα προϊόντα που αφορούν τις πρώτες ύλη μέσω ενός περιορισμού. Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Αρχή έκανε αναθεωρημένη πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη ε, τις δικές μας απαιτήσεις, ούτως ώστε να θέσουμε τα κατάλληλα όρια για κάθε είδους ε, προϊόν, θέλουμε να αξιολογήσουμε την πρόταση της αρμόδιας αρχής, να δούμε πώς το αναθεωρημένο καθεστώς καλύπτει τις υπερβολικές αλλαγές τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, διατηρώντας όμως και την αναγκαία Και για μη χρηματοστικές εταιρείε θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες είναι κατάλληλοι, και δεν θα ισχύουν για εκείνους που χρησιμοποιούν με υπεύθυνο τρόπο τι χρηματοπιστωτικέ αγορές για να μειώσουν το κίνδυνο ή όπου η χρηματοπιστωτική χρηματοσυντικη επιχειρηση τους είναι, το χρηματοσυντικό κομμάτι είναι μικρό σε σχέση με το τζίρο τους. Τώρα για την εφαρμογή των μέτρων του επίπεδου 2, ναι είμαι το ταχύτερο δυνατό να κινηθώ σε αυτό το τομέα, ε, ναι, δέχομαι απόλυτα ότι δεν θέλουμε μια επιταγή εν λευκό. Ε, και βέβαια θα εξασφαλίσω ότι οι υπάλληλοι μου θα ενημερώνουν πλήρως τη διαπραγματική ομάδα για την επιτυγχανόμενη ε, πρόοδο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Επίτροπε. Ο εισηγητής, ο κύριος Φέρμπερ, έχει το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά ευχαριστώ, ευχαριστώ όλου όσοι έλαβαν μέρο στη συζήτηση. Θέλω να διευκρινίσω τα εξή, ωστόσο. Εγώ, ω εισηγητή, ποτέ δεν θα δεχόμουν αναβολή εάν το ζητούσε μόνο ο κλάδο. Εδώ το να λέτε ότι υποτασσόμεθα στις επιταγές ε, του κλάδου προσβάλλει και το σώμα και την κοινή γνώμη. Απλώς δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλιστούν οι τεχνικές υποδομές και οι υποθέσεις εκείνες που θα επέτρεπαν στις εθνικές εποπτικές αρχές να επιτελέσουν σωστά το έργο τους. Δεύτερον, στις δύο εκθέσεις που θα ψηφίσουμε αμέσως δεν έχουμε να κάνουμε με το θέμα των ορίων θέσεων στις προθεσμιακές συναλλαγές. Έχουμε να κάνουμε με μια ρυθμιστική τεχνική ε, περιγραφή προτύπων που ακόμα πρόκειται να γίνει σε συζήτηση και όπου έχουμε εμείς ως Κοινοβούλιο ξεκάθαρα ορίσει και δηλώσει τη θέση μας και περιμένουμε η Επιτροπή να εκπληρώσει το καθήκον της. Δεν πρόκειται για αυτό το ζήτημα. Και τρίτον, στις συζητήσεις, στα θέματα στα οποία μιλήσαμε, δεν ε, εκτελέσαμε καμία επιταγή ή επιθυμία του κλάδου. Δύο χρόνια τώρα και οι σκιώδεις και ο υποφαινόμενος μήνα με το μήνα συνομιλούμε και καθόμαστε στο τραπέζι των συζητήσεων με την Επιτροπή και την ΕΑΚΑ για να επιλύσουμε τα επιμέρους προβλήματα ένα προς ένα. Ό,τι μας είπε η ΑΚΑ, ό,τι μας είπε η Επιτροπή είναι απλούστατα το εξή, ότι δεν μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα που επισημάνθηκαν διότι δεν το επιτρέπει η οδηγία. Και γι' αυτό θελήσαμε να κάνουμε τι σχετικέ προσαρμογέ. Αυτό σας το λέω και για την οδηγία, για το προσπέκτου, ε, για το δελτίο το ενημερωτικό και για όλα τα υπόλοιπα. Πρόκειται για ρυθμίσει οι οποίε δεν μπορούσαν να γίνουν στη μύφη, θα γίνουν μέσα στο στην νομοθεσία για το προσπέκτους και δεν έχουν καμία σχέση με τις επιθυμίες του κλάδου αλλά με ανάγκη για τεχνική προσαρμογή. Λοιπόν παρακαλώ να σταματήσουν αυτοί οι πενιγμοί ότι ανοίγει νέα παραθυράκια και πίσω πόρτες ο κλάδος προκειμένου να επιβάλλει τη δική του, το δικό του συμφέρον και τις επιθυμίες. Κατά τα άλλα ευχαριστώ όλους όσοι συνεργαστήκαν μαζί μου και αυτή η υποστήριξη μου δίνει θάρρος για να συνεχίσω και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την κατανόησή σας.